Um, good afternoon, ladies and uh, uh, Σας καλωσορίζω, σας ζητώ να δεχθείτε την μερίσια διάταξη. Έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί για την ψηφοφορία. Δεν την έχετε. Λοιπόν, όσοι την έχουν μαζί τους, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη. Να ζητήσω συγγνώμη. Ο πρόεδρος μας είναι στη Ουάσιγκτον με τον Διατλαντικό Διάλογο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος είναι επίσης απόν και θα προεδρεύσω εγώ εφόσον συμφωνείτε. Και είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε γιατί επιλογή δεν έχετε. να πω ότι το άρθρο 7, η αντιπροσωπεία του Χόκ στο Ζάγκρεμπ, δεν θα γίνει. Και η συζήτηση για τις δημόσιες προμήθειες που είχε προβλεφθεί για τις 10 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί σήμερα. Το πρόγραμμα για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες για το 2010 θα συζητηθεί επίσης. Πήρατε μια επιστολή όλοι από τη γραμματεία. Πρέπει κάπου να καταλήξουμε σήμερα. Συνεπώς η μερίσια διάταξη μπορεί να θεωρηθεί δεκτή. Σημείο 2. Ανακοινώσεις Προέδρου. Όλες οι επιστολές που ελήφθησαν μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνονται στους φακέλους σας. Για τα συμφέροντα των μελών οι επιστολές και ερωτήσεις γενικά πρέπει να ε, στραφούν προς τη γραμματεία. Να σας ενημερώσω ότι εκτός από το τμήμα και κλεισμένο των θυρών θα υπάρξει αναμετάδοση της συνεδρίασής μας. Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση, συνάδελφοι, στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, που διευρύνει τις αρμοδιότητές μας. Πρέπει να είμαι επιφυλακτικός αυτά που λέω, γιατί το κόμμα μου θα διαφωνεί με αυτά που λέω λίγον αλλά μιας και ομιλώ σαν πρόεδρος θα δείξουν κατανόηση. Είναι ευτυχής η ημέρα που συνεδριάζουμε λοιπόν στα πλαίσια της νέας συνθήκης και έχουμε πλέον συνομοθετικές αρμοδιότητες και για τα εμπορικά θέματα. Είναι ένα νέο κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι για την Επιτροπή μας ειδικά στο μέλλον προμηνύεται να είναι πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις αρμοδιότητές μας. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει λίγο περισσότερο το πώς βλέπει ότι θα αλλάξει ο τρόπος εργασίας μας. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά. Στο τέλος της συνεδρίασης θα γίνουν δεκτά. Αν έχετε ερωτήσεις λοιπόν για τα πρακτικά, να τις θέσετε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή τώρα για συγκεκριμένη ερώτηση. Όπως είπα στην αρχή της συνεδρίασης, παρακαλώ να έχετε τις κάρτες μαζί σας. Ελπίζω να έχουμε χρόνο. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4, δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας ΟΚΑΚΕ, συμφωνία Κοτονού. Δεν ξέρω, ο εισηγητής θα ήθελε κάτι να προσθέσει πριν την ψηφοφορία. Ναι ίσως και να μην είναι εδώ. Κάποιοι σκιώδεις εισηγητές θα ήθελαν το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε. Παράγραφος 1, τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν γίνεται δεκτή. Παράγραφος 2, τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 3. Δεν έχει καταπέσει, γιατί δεν έγινε δεκτή 2, οπότε την ψηφίζουμε λοιπόν. Την τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απολύπτεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 4. Η πέμπτη θα συνδυαστεί με το 4. Κατά. Δεκτή. Η πέμπτη θα συγχωνευτεί με την 4. Ποιοι είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Προφορική τροπολογία. Έχει κάποιος αντίρρηση για την προφορική. Θέλετε να τη διαβάσετε, Ντάνιελ, ή επειδή την έχουν όλοι μπροστά τους μπορούμε να προχωρήσουμε. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική του ΕΛΚ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 6 καταπίπτει. 7. Έτοιμα από τους σοσιαλιστές για τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεύτερο τμήμα. Απερίφθη το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτό. Παράγραφος 6. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξέχασα για τις αποχές μέχρι τώρα. Δεν μίλησα καθόλου για αποχές αλλά δεν τις ζήτησε και κανείς. Απερίφθη. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Εγώ ψηφίσω υπέρ, δεν έχω κάρτα σημειώστε το. 11 σημεία, 12 υπέρ δηλαδή. Τρεις αποχές, 12 υπέρ. Λοιπόν, 12 ψήφοι, 9 υπέρ, 2 αποχές. Λοιπόν, 10 υπέρ, 2 κατά, συγγνώμη για τη σύγχυση. Επόμενη ψήφος. Α, όχι, δεν υπάρχει επόμενη ψήφος. Περνάμε στο 5. Μέσα αμυντικά μέσα εμπορίου. Η αντιτάμπινγκ μέτρα. Cases. The main case which has been brought to the attention of our committee is the review. Λοιπόν, επανεξέταση τελών αντι-dumping για ορισμένα υποδήματα από το Βιετνάμ και την Κίνα. In Τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν στην Επιτροπή μας μετά από την απόφαση για επιβολή δασμών το 2006 στείλαμε επιστολές προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή επανειλημμένα ζητώντας την αναθεώρηση των μέτρων αυτών των οποίων η διάρκεια ήταν εκτάκτως περιορισμένη σε δύο έτη. Υπήρξαν αντιτιθέμενες απόψεις στη συζήτηση από το 2006 μέχρι τώρα. με την θέση σε ισχύ της συνθήκης, ίσως τα μέσα αυτά, εμπορικά μέσα άμυνας, να πρέπει να γίνουν πλέον διαφανή και να μην αντιτίθενται στα συμφέροντα των κρατών μελών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαλλαγεί της, των νέων ευθυνών του, αρμοδιοτήτων του, αλλά θα πρέπει να τις χρησιμοποιεί με αρελιστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα έχουμε στο μέλλον την δυνατότητα συζήτησης αυτών των νέων εμπορικών μέσων άμυνας θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει στάση και το ταχύτερο δυνατόν να ενημερώσει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλα τα μη επιχειρηματικά απόρριτα έγγραφα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μεταξύ των κρατών μελών μέσω της Επιτροπής Ad για την περίπτωση των υποδημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια πλήρη και κατανοητή παρουσίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης και των συστημικών επιπτώσεών της στο μέλλον των συστημάτων άμυνας του εμπορίου της Ένωσης. Όλοι είναι αλήθεια και σταματάει να διαβάζει ο κύριο Στέρντι. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό στο παρελθόν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, εγώ πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Προφανώς και τα συμφέροντα των κρατών μελών έχουν κυριαρχήσει πολλές φορές των μέσων άμυνας, αλλά ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια πλήρη παρουσίαση των θεμάτων και των θέσεων των κρατών μελών, εάν αυτό είναι εφικτό. Τον λόγο έχει πλέον ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντιπρέ. Ευχαριστώ. Το θέμα των υποδημάτων ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο, όπως γνωρίζετε. Και ήδη έχουμε το χρονοδιάγραμμα της αρχικής έρευνας για το αντι-dumping Πρόσφατα είχαμε την αναθεώρηση της ρήτρας εκπνοής. Δηλαδή τα μέτρα που είχαν υποβληθεί μια και εκπνέουν θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο θα παραταθούν ή όχι. Έγινε ενδελεχής έρευνα της υπόθεσης αυτής προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της. Δηλαδή κατά πόσο υπήρξε dumping, κατά πόσο εμπίπτει αυτό στον κανονισμό, αν συνεχίστηκε αυτή η πρακτική dumping. Uh, uh, uh, κατά πόσο υπήρξε βλάβη και αν συνεχίστηκε αυτή η οικονομική βλάβη. Εξετάσαμε όλες τις πτυχές ε, των κοινοτικών συμφερόντων και σχολιάσαμε τα πορίσματα της έρευνάς μας. Συντάξαμε ένα έγγραφο 86 σελίδων. Δεν χρειάζεται να το ανατρέξω λεπτομερώς. Πάντως τα βασικά μας πορίσματα είναι ότι από κάθε άποψη κρίναμε ότι υπήρξε συνέχιση των πρακτικών, ε, των πρακτικών dumping και πολλά μέτρα ε, που καλύπτονται από τη Συμφωνία Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και που στοιχειοθετούν πρακτική dumping. Και η μέθοδοι αυτή, η μέθοδος άλλες χώρες για παράδειγμα, αλλά και άλλοι δείκτες που εξετάστηκαν, όπως και να εξετάσαμε την υπόθεση, κρίναμε ότι υπήρξε και dumping και συνέχιση αυτής της πρακτικής. Τώρα το θέμα της βλάβης διαπιστώσαμε ότι το ντάμπινγκ των εισαγωγών είχε επιβλαβές αποτέλεσμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και επίσης διαπιστώσαμε ότι η βιομηχανία αυτή προσπάθησε να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να αντιμετωπίσει αυτές τις πρακτικές dumping παρά τη συνέχιση τους κατάφερε να επιβιώσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τα απορίσματα λοιπόν της ερευνάς μας προτείνουν συνέχιση των μέτρων anti-dumping για μία ακόμη περίοδο. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, κατά την οποία θα παραταθούν αυτά τα μέτρα anti-dumping, εξετάσαμε ποια είναι η κατάλληλη διάρκεια και με βάση τη διαδικασία και προσαρμογή εγκληματισμού της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας κρίναμε ότι μια παράταση κατά 15 μήνες αρκεί. Πριν βέβαια την ε, επανεισαγωγή, την επιβεβαίωση μέτρων, θα πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις τους σε άλλους οικονομικούς τελεστές και ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να διαπιστωθεί δηλαδή κατά πόσο τα μέτρα αυτά έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα σε άλλους οικονομικούς τελεστές ή στους καταναλωτές ενδεχομένω. Διαπιστώθηκε στην περίπτωση αυτή ότι τα μέτρα είχαν ελάχιστα σχεδόν μηδαμινά αποτελέσματα για τους ε, καταναλωτές μια και οι τιμές καταναλωτή προσδιορίζονται με πολύ διαφορετική βάση από ότι την τιμή προέλευσης, ε, στην προέλευση αυτών των προϊόντων. Οπότε από άποψη προστασία καταναλωτή δεν υπήρχε αντένδειξη για την θέσπιση, μάλλον την επανεισαγωγή των νέων μέτρων. Γι' αυτό και προτείναμε παράτασή τους για μία ακόμη περίοδο. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για την παράταση αυτή. Γι' αυτό και συνεχίζεται η διαδικασία επανεπιβεβαίωσης των μέτρων προκειμένου να επισημοποιηθεί αυτή η παράταση. Αν έχετε ε, απορίες συγκεκριμένε να σα απαντήσω. Πάντως είναι πολύ σύνθετη αυτή η υπόθεση. Θα μπορούσαμε να τη συζητούμε μέρες και εβδομάδες ολόκληρες. Θέλει κανείς το λόγο, υπάρχουν ερωτήσεις. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτό το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής ε, για το άρθρο 133. Θα ήθελα να, μου πείτε ποιο αποτέλεσμα προέκυψε τελικά από τη συναντήση αυτή και πώς θα συνεχίσει τις εργασίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, γιατί κάποια κράτη-μέλη προτιμούν να διατηρηθούν οι δασμοί αυτοί και τι θα κάνει λοιπόν η Επιτροπή στα πλαίσια της Επιτροπής 100, του άρθρου 133 και θα δεθεί αυτό το θέμα επί της αρχής γιατί το... η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχει κάποια επιρροή, κάποια επίδραση και σε ό,τι αφορά τα μέτρα εμπορικής άμυνας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενταχθούν και τέτοια μέτρα στα πλαίσια της ε, αντιμετώπισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήσει και το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στο μέλλον για τέτοια μέτρα anti-dumping. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα μέτρα anti-dumping και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να απαντήσει την ερώτηση του Ντάνιελ. Στην περίπτωση αυτή των υποδημάτων ή τις ευρύτερες επιπτώσεις της, εμείς προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυστηρά τους κανόνες και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον κατά τη γνώμη μου. Θεσπίσαμε ένα πλαίσιο στο βασικό κανονισμό που προβλέπει την ακολουθητέα διαδικασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου συγκρούνται διάφορα συμφέροντα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο τεχνικοί και επαγγελματικοί γίνεται και να προβούμε, να προβούμε σε μια πολύ ρεαλιστική ανάλυση. Βέβαια είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και έγινε διάφορα πάθη αριστερά και δεξιά αλλά τα κράτη-μέλη τελικά επιβεβαίωσαν ότι ο καταλληλότερος τρόπος ε, προσέγγισης τέτοιων υποθέσεων είναι να είμαστε όσο πιο τεχνικοί γίνεται και να τηρήσουμε τις παραμέτρους του κανονισμού. Μάλιστα έρχομαστε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάζουμε τέτοιες υποθέσεις και όπως προτείνετε κι εσείς ε, θα το πράξουμε και στο μέλλον. Μας ενδιαφέρει αυτή η ανταλλαγή απόψε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις, για ε, τις υπόλοιπες αποφάσεις αποτελούν τμήμα μιας γενικότερης διαδικασίας στα πλαίσια της επιτροπολογίας ή των αποφάσεων της διαδικασίας επιτροπολογίας. Και είναι και το κατάλληλο πλαίσιο για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Ελπίζω να σας ικανοποιήσει η απάντηση. Άλλος κανείς? Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από το κρατήριο, θα ήθελα και εγώ να θέσω ορισμένες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γερμανία, η Μάλτα και η Αυστρία αποφάσισαν στον προηγούμενο γύρο να απέχουν στην τελευταία ψηφοφορία, παρά να εξακολουθούν να θίστανται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει γιατί επαναχώρησαν αυτές οι τρεις χώρες στην συνεδρίαση την τελευταία γιατί από ό,τι ξέρω, και ίσως το γνωρίζει καλύτερο ο Ντάνιελ, οι Γερμανοί αποφάσισαν να πόσχουν μια και οι τελωνιακοί δεσμοί ούτως ή άλλως θα έλεγαν μέσα σε 15 μήνες, παρά το, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχουν νομικά εχέγγυα για κάτι τέτοιο. Μπορεί να επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβεβαίωση που έδειξε η Γερμανία και ποια είναι η νομική βάση τέτοιου είδους διαβεβαιώσεων. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο θέμα για τις επιπτώσεις στον καταναλωτή, το κόστος για τον καταναλωτή μετά την εισαγωγή αυτών των δασμών. Δεν πιστεύετε ότι πολλοί λιανέμποροι θα χρειαστεί να απορροφήσουν αυτό το κόστος και να το εντάξουν στη διαδικασία προμήθειας και παραγωγής. Και μάλιστα μεσούς της χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν ξέρω αν είναι καλή αυτή η εξέλιξη. Πολύ φοβούμαι ότι δεν θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ε, ευρωπαϊκής υποδηματοποίησης με τέτοιου είδους δασμούς. Και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το κόστος δεν έχει αυξηθεί, θα έχει πολύ λίγο χρόνο η Ευρωπαϊκή Υποδηματοποίηση για να απορροφήσει αυτό το επιπλέον κόστος. Γιατί αν συνεχίσει να το απορροφά για πολύ χρόνο, τότε δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν η Γερμανία, η Ευστρία και η Μάλτα άλλαξαν άποψη. Ίσως να πίστηκαν από τις προτάσεις μας. Αρχικά, θέλανε απλά να έχουν πιο πολλά επιχειρήματα, πιο πολλές ε, πιο πολλά προδεικτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι τελικά τους πείσαμε και έτσι αναθεώρησαν τις τάσεις τους. Γιατί στην Επιτροπή πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτή ήταν η σωστή στάση και εξηγήσαμε εις την περίπτωση αυτή. Κάποια στοιχεία, ωστόσο, δεν διευκρινίστηκαν απόλυτα για κάποιους, μέχρι σε και πολύ ύστερη φάση στις διαπραγματεύσεις. Ένα από τα στοιχεία τα οποία δεν ήταν σαφές για τα κράτη-μέλη ήταν ότι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη συγκρισιμότητα των προϊόντων, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε πραγματικά αποτεκτικά στοιχεία. Είχαμε ήδη σημειώσει ότι τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα, αλλά νομίζω ότι χρειάστηκαν τελικά κάποια αποτεκτικά στοιχεία χειροπιαστά για τη συγκρισιμότητα των προϊόντων, τα οποία τα είδαμε πολύ μετά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο και καθόρισε την στάση των χωρών αυτών εν τέλει. Επίσης, για παράδειγμα, η Γερμανία θεώρησε ότι καλό θα ήταν η ευρωπαϊκή βιομηχανία να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να προσαρμοστεί και ήθελε κάποιες διευκρινήσεις για την ταχύτητα της ε, προσαρμογής αυτής. Φυσικά αυτό χρειάστηκε να το μελετήσουμε, να το ερευνήσουμε και τα αποτελέσματα τα είδαμε σε μετέπειτα φάση. Και έτσι λοιπόν κατέληξαν στα συμπεράσματά τους τα κράτη-μέλη, γιατί τελικά πίστηκαν ότι είχε ξεκινήσει μια σωστή διαδικασία προσαρμογής. Σε ό,τι αφορά το θέμα του αντικτύπου για τον καταναλωτή και σε ό,τι αφορά το κόστος. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε ή ήταν τον αντικτύπωση που υπήρξε για τον καταναλωτή. Και αυτό εξηγείται σε διάφορα έγγραφα. Εισαγωγής κυρίως, υπέστησαν κάποιες οικονομικές ε, συνέπειες σε ό,τι αφορά τους δασμούς αυτούς. αλλά εξετάσαμε προσεκτικά, και αυτό αποτελεί τμήμα της αποναμαζόμενης ε, κοινωτικής ανάλυσης, κατά πόσο αυτό θα διακύβευε το έργο των εισαγωγέων. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι ναι δεν υπήρχαν κάποια, κάποιες οικονομικές ε, συνέπειες, αλλά παρ' αυτά το περιθώριο κέρδους των εισαγωγέων ήταν ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά την παράταση των μέτρων αυτών και ότι δεν ε, υπήρχε κανένας κίνδυνος να υποστούν νέες ε, ζημιές εισαγωγής. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κοιτώντα το θέμα των εισαγωγών υποδημάτων προς την Ένωση, τα προϊόντα ε, αντιπροσωπεύουν το 7% περίπου της συνολικής αγοράς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αρνητικές συνέπειες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό ειλικρινά θα διακύβευε τη θέση των εισαγωγέων. Σε ό,τι αφορά τους λιανέμπορους τώρα, μπορεί οι εισαγωγείς ε, να είχαν ασκήσει όντως κάποια πίεση στους λιανέμπορους για να αναλάβουν τμήμα του απολεσθέντος κέρδους. Ωστόσο, και πάλι διαπιστώνουμε ότι το 93% όλων των υποτιμάτων, δεν υφίσταται, δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα αυτά. Άρα, εξετάζοντας την κατάσταση των λιανεμπόρων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για ένα μικρό τμήμα μόνο της συνολικής τους, ε, του συνολικού τους εμπορεύματος. Και επίσης, οι λιανέμποροι δεσμεύονται και από τον, την τοποθεσία της πώληση. Γιατί Μπορεί να φανταστούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μετεγκατάστασης σε χοντρικό επίπεδο, αλλά σε λιανικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια μετεγκατάσταση. Uh, I think Ναι, όντως, απίθανο. Ο Ντάνιελ. Ναι, για να μην έχουμε εδώ πέρα παρεξηγήσεις, νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό το γεγονός ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρατείνει του τελενιακού δασμού, αλλά θέλω να ξέρω το εξή. Εφόσον τέθηκε λοιπόν πλέον σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, από ό,τι καταλαβαίνω η νομική πραγματικότητα ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πράξη για να επικρατήσουν τα μέτρα αυτά. Ισχύει αυτό ή μπορεί να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά βάσει της παλιάς ε, ε, νομικής βάσης, γιατί αν ισχύει κάποια στιγμή θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τέτοια έγκριση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο. Και αυτό δεν έχει συμβεί τις τελευταίες, τις τελευταίες 7 ημέρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω επί ποιας νομικής βάσης θα αριστούν τα μέτρα αυτά είναι εδώ και οι νομικές υπηρεσίες, αλλά μήπως θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Ε, μια και είναι εδώ η νομική υπηρεσία, προτιμώ εκείνη να απαντήσει. Ah, yeah, um, we have actually... Έχουμε ήδη απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ο κανονισμός που ισχύει από το 1996 συνεχίζεται κανονικά και μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κανονισμός αυτός δεν μπορεί να αλλάξει και αν αλλάξει. Αυτό θα πρέπει να γίνει από την κανονική νομοθετική διαδικασία και το Κοινοβούλιο σα συνομοθέτει. Μέχρι ότου να γίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον κανονισμό ως έχει. Οι μεμονωμένες αποφάσεις για το anti-dumping θα συνεχίσουν να λαμβάνονται δηλαδή προς το παρόν από το Συμβούλιο. Αυτό απαντά την ερώτησή μου για την κατάσταση στη Γερμανία. Διερωτώ με πώς θα πάρει τις εγγυήσεις που θέλει η Γερμανία ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ζητήσει και θα αποφασιστούν από το Συμβούλιο και θα υπάρξει συμφωνία μάλλον στο Συμβούλιο για να τερματιστεί η επιβολή των μέτρων αυτών μετά από 15 μήνες. Δεν ξέρω αν θα ζητήσουν μια ποσοτική απάντηση. Αν θέλουμε να αποφασίσουν λοιπόν για μέτρα που θα διαρκούν 15 μήνες, αυτό θα το αποφασίσει το Συμβούλιο η απόφαση που επιβάλλει τα μέτρα είναι απόφαση του Συμβουλίου. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Στέφαν. Πήρε μέρος σε κάποιες συναντήσεις τις οποίες είχαμε μη πολιτικής φύσης, ιδιωτικές πολλές φορές, για να κατανοήσουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν είναι και αυτός τόσο υπέρμαχος της απόλυτα ελεύθερης αγοράς, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει να συζητάμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τα της Λισαβόνας, θα συνεχίσει να είναι δεκτική απέναντί μας και να συνεχίσει να μας ενημερώνει για τους τρόπους και λόγους μάλλον για τους οποίους λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Το επόμενο είναι το 6. Αντιπροσωπεία της ΣΥΝΤΑ Μαδλώνα, τη Μαδρίτη. Όχι για τις σταυρομαχίε. Πριν από την Ισπανική αντιπροσωπεία είχαμε συζητήσεις ε, με εκπροσώπους της κυβέρνησης για τα θέματα του εμπορίου και συζητήσαμε με εταιρείε εξαγωγικές προς τον τρίτο κόσμο. Ο κύριος Κάζακ ήταν ο υπεύθυνο της αντιπροσωπείας, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ, μέλος της Επιτροπής σας έτσι κι Θα ακούσουμε με ενδιαφέρον αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφε. Όπως είπατε, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας Διεθνούς Εμπορίου πήγε στην Ισπανία, όχι μόνο στην Παμπλώνα, αλλά και στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε εκπροσώπους της τοπικής κυβέρνησης της Ναβάρας και επίσης υπουργού και γενικούς γραμματείς υπουργείων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για θέματα διεθνούς εμπορίου. Συναντηθήκαμε επίσης κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς μας στην Αβάρα με δύο από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα την Παμπλώνα και οι οποίες εξειδικεύονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίσκεψη αυτή είχε σαν στόχο την αποκοινού εξέταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια και της επερχόμενης Ισπανικής Προεδρίας γύρω από το διεθνές εμπόριο. Νομίζω ότι η Προεδρία αυτή όλοι υπογράμμισαν ότι ε, καλείται να αναλάβει σε μια κρίσιμη στιγμή μετά την εισαγωγή της συνθήκης και μετά από την αναβάθμιση του ρόλου που, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της δικής μας Επιτροπής για τη σωστή άσκηση της ε, εξωτερικής εμπορικής πολιτικής. Αυτό υπογραμμίστηκε και στις επαφές τις οποίες είχαμε με τον πρόεδρο της τοπικής βουλής, με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και με τον Υπουργό για το Διεθνές Εμπόριο της κυβέρνησης της Μαδρίτης και με τον Υφυπουργό για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανική Προεδρία είναι ιδιαίτερος φιλόδοξη. Σκοπεύει να αντιμετωπίσει με πολλή ενέργεια θα έλεγα όλες τις εκκρεμότητες οι οποίες έχουν σωρευτεί τον τελευταίο καιρό και απαιτούν μια ιδιαίτερα δραστήρια αντιμετώπιση. Έγινε αναφορά στον κύκλο της Ντόχα, έγινε αναφορά επίσης στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με διάφορες χώρες. Ε, θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά και στις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής εδώ από τους Ισπανούς, όπως επίσης και για την Ευρωμεσογειακή Ένωση. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουν σαν στόχο να καταστήσουν το διεθνές εμπόριο απαραίτητο μέσο καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης και οικονομικής αηφόρου ανάπτυξης κάτι που με τη σειρά του θα επιτρέψει την βελτίωση των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση στη Ναβάρα, είναι όταν είδαμε ότι στα πλαίσια της συνάντησης κορυφής της Κοπενχάγης για τις κλιματολογικές αλλαγές η περιοχή της Ναβάρα η περιφέρεια της Ναβάρα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα για τις ανανεώσιμες πηγές. Ήρθαμε σε επαφή με την Αξιώνα Ενέργεια και την Εμτορές. Η Αξιώνα Ενεργεία είναι ηγέτης παγκόσμια στα ε, αιωλικά. Έχουν εγκαταστήσει άνω των 200 αιωλικών εγκαταστάσεων στον κόσμο και η περιφέρεια της Ναβάρα συνεπώς έχει πετύχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα γιατί το 50% της ενέργειας της περιφέρειας της Ναβάρα προέρχονται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Συζητήσαμε επίσης για τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι ισπανικές και ευρωπαϊκές τεχνικές εταιρείες όταν έρχονται σε εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και συζητήσαμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την απόσυρση όλων των εμποδίων στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η επίσκεψη λοιπόν νομίζω ότι ήταν πολλαπλά ενδιαφέρουσα για μας όλους και περιμένουμε με ανυπομονησία την συνάντηση την οποία θα έχουμε στις αρχές του επομένου έτους εδώ στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Εμπορίου της Ισπανίας και με τους Ισπανούς εκπροσώπους για να δούμε με ποιο τρόπο στα πλαίσια της εφαρμογής της συνθήκης η φιλόδοξη αυτή στόχη οι οποίοι θα ποσοστικοποιηθούν από την Ισπανική Προεδρία θα γίνουν αντικείμενο, θα, γενικά θα πετύχει η Ισπανική Προεδρία στους στόχους που θα θέσει. Ευχαριστώ και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που έχουν προετοιμάσει ε, κάποια σημαντικά μνημόνια γύρω από τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας. Αν θέλετε κάποια συμπληρωματική πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Καζάκ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Σας ευχαριστώ που ήσταν επικεφαλής αντιπροσωπείας που αν δεν κάνω λάθος ήταν επιταμελής. Και ήταν πολύ επιτυχημένη αυτή η αντιπροσωπεία γιατί συνήθως ε, δηλώνουν υποψηφιότητες πολλά μέλη αλλά δεν πηγαίνουν στις αποστολές. Τελευταία φορά είχα πάει πριν από 48 χρόνια ε, ε, για το έθιμο αυτό των τάβρων στην Παπλώνα. Και σίγουρα πολλά θα έχουν αλλάξει. Σήμερα δεν θα είχα το κουράγιο να το κάνω. Πάντως ε, δίκιο έχετε ότι η Ισπανική Προεδρία θα αναλάβει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Προεδρία της. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος το λόγο ή κανένα άλλος που ήταν παρόν στην αντιπροσωπεία να λάβει το λόγο. Όχι. Κανεί από την αντιπροσωπεία δεν είναι εδώ εκτό από τον κύριο Καζάκ. Σα ευχαριστούμε θερμά. Πάντω, όντω, ε, στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία αυτή η αποστολή. Σημείο 7. Είπα στην αρχή ότι η αντιπροσωπεία του Χόκ στο Ζάγκρεπ ε, Κροατία μεταφέρθηκε, αναβλήθηκε για την επόμενη μας συνεδρία στις 10 Δεκεμβρίου. Επόμενο θέμα είναι οι δημόσιες προμήθειες. Είναι συνεχής ε, ο αγώνας και σφοδρές συζητήσεις για το θέμα των δημοσίων προμηθειών και από τότε που ασχολούμαι με το διεθνές εμπόριο ανέκαθεν ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά των δημοσίων προμηθειών και της έλλειψης πρόσβεσης ορισμένων εταιριών στις αγορές χωρών που είναι κοντά μας και έχουν τεράστιο δυναμικό και ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μάλιστα, η αγορά αυτή είναι 60% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Τεράστια σημασία δηλαδή. Μάλιστα, η Επιτροπή ΕΜΚΟ ετοιμάζει έκθεση της πρωτοβουλίας για τις εξελίξεις στις δημόσιες προμήθειες και πολύ σημαντική οικονομική εταίρη υιοθετούν ε, περιοριστικές πρακτικές πρόσβασης στις δημόσιες προήθειες. Είναι ένα είδος ε, μέσω εμπορικής άμυνας και είτε αποκλίνω από την αρχή από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή ε, συμμετέχουν αλλά με δυσμενέστερες προϋποθέσεις από ό,τι οι ντόπιοι ανταγωνιστές. Θέλουμε να ανοίξει αυτή η αγορά δημοσίων προμηθειών στον κόσμο και να φροντίσουμε ότι και η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει αθέμητη εκμετάλλευση της ε, εσωτερικής αγοράς από τρίτες χώρες. Θα πρέπει το θεμητό εμπόριο και οι δημόσιες προμήθειες να γίνονται με πνεύμα αμοιβαιότητας. Δεν ξέρω ποιος ε, θα λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ο μιλητής προβλεπόμενος. Α, ο εισηγητής καταρχήν. Να σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Χάντζλικ. Μπορώ να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτά τα θέματα δημοσίων προμηθειών έχουν τεράστια σημασία για την οικονομία και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο υπενθυμίζω αυτό που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι οι δημόσιες προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου το 60% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οπότε το άνοιγμα των δημοσίων προμηθειών στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς θα αυξήσει, αυξάνει, τον ανταγωνισμό και δημιουργεί πολλές οικονομίες. Αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη όλες οι ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς για τις δημόσιες προμήθειες. Πολλά θα πρέπει να μείνουν ακόμη. Επίσης, πολλά θα πρέπει να γίνουν σε θέματα διεθνούς συνεργασίας. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι η προσέγγιση αυτή, την προσέγγιση αυτή μάλλον δεν την εστερνίζονται οι διεθνείς μας εταίροι. Γιατί οι κύριοι εμπορικοί και οικονομικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν περιοριστικές πρακτικές στα θέματα δημοσίων προμηθειών, που είναι πολύ πιο ορατές σήμερα εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης οι δημόσιες προμήθειες είναι για τους εξαγωγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μια, ένα πεδίο ανεκμετάλλευτων ευκαιριών. Και οι επιχειρηματίε Ένωση έχουν κορυφαία θέση σε πολλού τομεί, αλλά εξαιτία των περιοριστικών πρακτικών δημοσίων προμηθειών δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ε, σημαντική του θέση. Και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι μεσαίοι επιχειρηματίε έχουν τεράστιο δυναμικό καινοτομία, ιδιαίτερα στις, ε, τους τομείς που είναι και νης τομείς αριστείας και δυστυχώς προσκρούν σε αρνητικές κυβερνητικές πρακτικές των τρίτων χωρών και περιοριστικές και ακόμη και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου βρίσκεται υπό αναθεώρηση σχετική συμφωνία. Περιμένουμε μια βελτίωση της κατάστασης για, τις, για τους επιχειρηματίες μας. Το καλύτερο θα ήταν να υλοποιηθεί συμφωνία την οποία όμως θα προσυπογράψουν όλες οι χώρες ή τουλάχιστον οι περισσότερες χώρες που είναι μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Γιατί αυτή τη στιγμή συμβαλόμενα μέρη της συμφωνίας είναι κυρίως ε, ε, ανεπτυγμένες χώρες. Βέβαια σε μακροπρόθεσμη προοπτική αυτή είναι και η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μα δώσει κάποιε πληροφορίε ε, για την κατάσταση των ε, εργασιών και τι εξελίξει ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη συμφωνία για τι δημόσιε προμήθειε στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Φυσικά γίνονται διμερείς διαπραγματεύσεις και με χώρες για τις δημόσιες προμήθειες. Πολλές φορές έχουμε συμβάσεις ελευθερού εμπορίου με τη Χίλη και το Μεξικό, για παράδειγμα, ή με το Κάριφόρ. Ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι οι νέε ε, εμπορικές συμφωνίες, ε, που θα είναι το νέο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής, θα καλύπτουν και την περίπτωση των δημοσίων προμηθειών. Περιμένω όμως την παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να μας πει πώς και σε ποιο βαθμό η υποδιαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν υπόψη και το θέμα των δημοσίων προμηθειών, στα θέματα της εσωτερικής αγοράς ή τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κάποια κοινωνικά ζητήματα. Και τέλος, ε, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα. Η γνωμοδότηση θα υποβληθεί μέχρι τις 8 ή το αργότερο 11 Ιανουαρίου, τότε που θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, στις 27 θα το συζητήσουμε και στις 29 λίγη προθεσμία, 29 πρώτου για τις τροπολογίες, ενώ στις 23 Φεβρουαρίου προβλέπεται η συζήτηση στην Επιτροπή μας. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα, 29 πρώτου η λίγη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και 23 Δευτέρου συζήτηση στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Uh, Ονομάζομαι Σπίγκελ από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Μονάδα Δημοσίων Προμηθειών. Η κυρία Ρίλε εκπονεί αυτή τη στιγμή την έκθεση της πρωτοβουλίας για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Γι' αυτό ήρθα και εγώ εδώ, γιατί από ό,τι ξέρω η έκθεση αυτή θα επικεντρωθεί σε πολλά σημεία της εσωτερικής αγοράς και εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίου προμηθειών εντός της εσωτερικής αγοράς. Η κυρία Ρίλη, η της ΣΥΜΚΟ, ανήγγειλε ότι θα επικεντρωθεί σε δύο κυρίως νομικά θέματα και νομικά προβλήματα. Τα θέματα σχέσεων στο δημόσιο και σε ό,τι αφορά τις, την υλοποίηση των στόχων Τη συνθήκη τη Λισαβόνα, πώ θα εφαρμοστούν αυτοί στα θέματα των δημοσίων προμηθειών. Επίση, ε, λέφθησαν υπόψη οι περιβαλλοντικέ δημόσιε προμήθειε καινοτόμε, κοινωνικέ, αηφόρες, δημόσιε προμήθειε, διάφορε πτυχέ. Και εγώ είμαι εδώ για να παρακολουθήσω τη συζήτηση για αυτά και να σα δώσω τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σημεία αυτά. Αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να σα ενημερώσω για τις εξελίξεις ε, των συζητήσεων σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Γιατί η αρμόδια για το θέμα αυτό είναι άλλη υπηρεσία. Πάντως θα διαβιβάσω στον αρμόδιο τις ερωτήσεις σας, ώστε να συμφωνήσετε μια παρουσίαση άλλη στιγμή. Κυρία Χάντζλικ, έχετε κάποιο σχόλιο? Καλώς, ε, πολύ σωστό να διαβιβάσετε στον αρμόδιο τις ερωτήσεις μου και αν μπορεί να απαντήσει είτε γραπτός είτε με άλλο τρόπο θα ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Yes, I agree there. Um, could I just ask uh, the Commission? Καλώς. Ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα μίλησε για την εσωτερική αγορά και την κατάσταση των δημοσίων προμηθειών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμω ότι ε, ότι η δική μας αγορά, η εσωτερική αγορά είναι σχετικά ανοιχτή σε θέματα δημοσίων προμηθειών. Τι θα γίνει, θα την ανοίξουμε ακόμη περισσότερο, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες μεγαλύτερου ανοίγματο. Γιατί είπατε ότι καλύπτεται μόνο την εσωτερική αγορά. Αλλά τι γίνεται με τη πρόσβασή μας στην αγορά δημοσίων προμηθειών τρίτων χωρών, έξω κοινοτικών χωρών. Όπως είπατε, οι δικέ μας αγορέ, η δική μας εταιρεία αγορά είναι σχετικά ανοιχτή για τις δημόσιες προμήθειες. Ιδιαίτερα για κρατικές προμήθειες, για κυβερνητικέ προμήθειε. Στις τρίτες χώρες βέβαια την απόφαση τη λαμβάνουν ε, μεμονωμένα θα ανοίξουν τις δημόσιες τους προμήθειες ή όχι. Και έγιναν πρόσφατα πολιτικές συζητήσει. για τη συμμετοχή κινέζικων εταιριών σε κάποια κατασκευαστικά έργα στα κράτη-μέλη. Αλλά τώρα, αυτή είναι η γενική κατάσταση. Υπάρχει συζήτηση για την διάβρεση του κύκλου των χωρών GPA με βάση συγκεκριμένες ειδικέ συμφωνίες. Για όλα αυτά θα σας ενημερώσει συνάδελφος από, την ομάδα που είναι, από τη μονάδα που είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά. Um, ναι, προτείναμε πριν από λίγο στην επόμενη συνεδρίαση ο αρμόδιος να είναι εδώ και αν θα μπορούσατε να έχετε επαφές την κυρία Χάντζλεκ. Ναι, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ προσωπικά καλύπτω την έκθεση Ρίνα και επειδή η έκθεση αυτή εστιάζεται σε θέματα εσωτερικής αγοράς, με έστειλαν για να καλύψω τα θέματα αυτά. Αλλά φυσικά θα φροντίσουμε προκειμένου να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που θέλετε. Ναι, ευχαριστώ, λέγε ο Πρόεδρος. Αυτό νομίζω ότι απασχολεί πολλούς βουλευτές. Γι' αυτό και το θέσαμε το θέμα. Γι' αυτό και η κυρία Χάντλικ θα φροντίσει να έλθει εδώ αρμόδιο στην επόμενη συνεδρίαση. Κάνει άλλο παρακαλώ. Να περάσουμε στο 8. Τρέχουσε εξέλιξει όσον αφορά συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία, ότι ένας από τους ε, εισηγητές που ασχολήθηκε την προηγούμενη θητεία με τα θέματα αυτά και έχουμε και τον David Martins εδώ που ασχολούνται με θέματα οικονομικών εμπορικών σχέσεων. Θεωρούμε ότι η παρούσα φάση αποτελεί εταιρική συμφωνία σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Και χάρη στη γραμματεία και στις δικές μου προσπάθειες, ε, γιατί προσκαλούμε εδώ και καιρό την γραμματεία, είναι σημαντικό το ότι έχουμε πετύχει συμφωνία σε μία από τις έξι διαπραγματευτικές ομάδες. Συμφώνησε το Κοινοβούλιο και το 2004 παρακολουθούμε τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές με διάφορες περιφέρειες και διοργανώθηκαν και και κλεισμένε συνεδριάσει με την Επιτροπή, αλλά και ανοιχτέ συνεδριάσει στο Κοινοβούλιο με την Κοινωνία των Πολιτών και το καθεξή διαβουλεύσει και αποτελεί μία από τι διαρκεί ε, δεσμεύσει τη Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες αυτές οι οικονομικές συμφωνίες και ε, ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ευχαριστώ. η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης Η τελευταία ενημέρωση έγινε ουσιαστικά τον Οκτώβριο του 2009 και αν δεν κάνω λάθος αυτό εστάλει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς ε, έχουμε φτάσει τώρα στις αρχές Δεκεμβρίου και θα ήθελα να δούμε ακριβώς τι έχει αλλάξει πρόσφατα. Υπάρχει το θέμα της Συμφωνίας Καμπίν, είναι η Συμφωνία ουσιαστικά η οποία αντιμετωπίζει σε περιφερειακό επίπεδο τα προβλήματα. Δεν έχει υπογράψει η ΑΕΤ ακόμα. Η ΑΕΤ μαθαίνουμε ότι προετοιμάζεται να υπογράψει σύντομα. θα γίνουν οι δασμολογικές προσαρμογές οι οποίες ζητήθηκαν από τη χώρα αυτή. Είναι μια θετική πρώτη κίνηση και επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση, θα επιβεβαιωθεί μάλλον στη συνάντηση κορυφής που θα γίνει το 2010, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί η ημερομηνία. Μια άλλη πληροφορία που έχω, ίσως να μην είναι κάτι το νέο για όλους, είναι ότι τα Φίτζι αποφάσισαν ότι θα υπογράψουν και αυτά, την ενδιάμεση είπα συμφωνία δηλαδή, το ίδιο έκανε και η PNG νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίε προς το παρόν, είναι θέμα πρακτικών ρυθμίσεων. Δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες ε, για τις υπόλοιπες ελίπουσες υπογραφές, την ε, Νότιο-Ανατολική Αφρική, Γκάνα, Ναμίμπια, Κομόρες και Ζάμπια. Να σας διαβεβαιώσω μόνο ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τις χώρες αυτές για να ε, προχωρήσουμε σύντομα. για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Να σταθώ λίγο στις διαπραγματεύσεις στη Δυτική Αφρική που έχουν προχωρήσει αρκετά. Είναι σαφές ότι παρά τις καλές προθέσεις όλων μας, η προθεσμία της 10ης Οκτωβρίου δεν έγινε σεβαστή και δεν θα τερματιστούν φέτος οι διαπραγματεύσεις αυτές. Ελπίζουμε όμως να ολοκληρωθούν το 2010. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, θα σταματήσω εδώ. Θα πω μόνο ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε τη συζήτηση γύρω από αυτές τις συμφωνίες, όχι μόνο σε αυτό το φόρουμ, αλλά με όλους τους εμπλεκομένους. Προγραμματίζονται κάποια σεμινάρια για αυτές τις συμφωνίες στις χώρες ΑΚΕ το 2010 για να προωθηθούν οι συγκεκριμένες αυτές μορφές συνεργασίας. Ευχαριστώ, Ντάνιελ. Ναι, μία ερώτηση μόνο να κάνω. Όταν γνωρίστηκε ο Επίτροπος διάβασα σε κάποιες εφημερίδες ότι ο Ντεχούχτ στο παρελθόν ασχολούταν με θέματα για τις ε, χώρες τις αναπτυσσόμενες. Άρα μπορεί να δίνονταν νέα όθηση στο θέμα των συμφωνιών ΙΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και ότι μάλλον η Βαρόνι Άστον δεν θα είχε κάνει τέτοιες, ε, δεν θα είχε αναλάβει τέτοιες δράσεις Ήθελα να σας ρωτήσω, τις τελευταίους έξι μήνες όντως δεν έχει κινηθεί τίποτα σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ΕΠΑ. Γιατί αν σωστά κατάλαβα αυτά που μας είπατε, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εξελίξεις, ιδιαίτερη πρόοδος. Υπάρχει κάτι το καινούργιο, γίνονται νέες διαπραγματεύσεις. Προβλέπετε κάτι για τη σύναψη νέων συμφωνίων ΕΠΑ ή απλά περιμένουμε να υπογραφούν όλες οι προσωρινές συμφωνίες ΕΠΑ. David. Όπως και ο Ντάνιλ, θα ήθελα και εγώ να συμφωνηθούν και να υπογραφούν οι συμφωνίες, ΕΠΑ. αλλά νομίζω ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή και θα ήθελα να ρωτήσω και να ζητήσω να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν ε, παρενοχλούμε ιδιαίτερα τις χώρες της Δυτικής ε, Αφρικής να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες. Ότι δηλαδή τους δίνουμε το χρόνο που χρειάζονται για να πληροφορηθούν, για να μάθουν τι είναι οι συμφωνίες ΕΙΠΑ, να μάθουν από τις ίδιες αυτές τις ε, συμφωνίες ΕΙΠΑ σε ό,τι αφορά την Καραϊδική. Ο Κάρλ Ντεχούχτη είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν ήθελε να σχολιάσει ιδιαίτερα το θέμα των ε, ΙΠΑ, των συμφωνιών ΙΠΑ. Και ότι θα το κοιτούσε το θέμα αυτό αργότερα, όταν θα διοριστεί η Επίτροπο Εμπορίου. Αλλά υπονόησε ότι δεν επρόκειτο να σπρώξει υπερβολικά τα πράγματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, όντω, όπως είπε και ο κύριος Μάρτιν, να πω δύο λόγια για το τι έγινε στη Ρουάντα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου έγινε μια συνάντηση ειδικά για τι συμφωνίε ΕΙΠΑ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και οι θέσει των συναδέλφων εκ μέρου των χωρών ΑΚΕ. Επειδή η συνάντηση έλαβε χώρα στην Ρουάντα, μια χώρα με τις πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Δυτική Αφρική, Η Σαντέκ έχει υπογράψει τις συνθήκες της συμφωνίας, είπα, αλλά όχι η Αγγόλα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία υπάγεται στο Σαντέκ, αλλά η ίδια η χώρα αυτή δεν έχει υπογράψει τις συμφωνίες, είπα. Μόνο οι πιο μικρές ε, χώρες έχουν υπογράψει το Λεσότο, η Σουαζιλάνθη και η Μποτσιγάνα. Και νομίζω και η Μοζαμβική ίσως. Στην αρχή λοιπόν της συνάντησης ε, ο συμπρόεδρος Ράσμουσεν είπε ότι είναι πολύ δύσκολο για μας ε, να συνάψουμε τις συμφωνίες αυτές ΑΚΕ, είπα συγγνώμη, γιατί τα προϊόντα μας δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τοπικά τα τοπικά προϊόντα και χρειαζόμαστε την εμπορική υποστήριξη και την υποστήριξη marketing εκ μέρους της Ευρώπης προκειμένου να αποδεχτούμε τα νέα αυτά σχέδια. Και την τελευταία φορά που παρευρέθηκα στη Γενέβη για την ε, εκτελεστική επιτροπή, συνάδελφοι από την Αμίμπια παραπονέθηκαν σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην αγορά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα πλέον είναι πιο φτηνά από τα προϊόντα της Ναμίμπια. Και αυτό αποτελεί απόρρια των εξαγωγικών ενισχύσεων εκ μέρους μας. Αυτά για να σας πω ότι δεν με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα σχόλια του Διευθυντή Τόμψον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρευρέθηκε. Δεν υπάρχει μια σαφή στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και με απασχολεί το τι θα γίνει με τις συμφωνίες, είπα. Αλλά προφανώς θα πρέπει να κινηθούμε προς τρεις κατευθύνσεις. Καταρχάς, να είναι δυνατή η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνονται πολύ πιο πολλές διαβουλεύσεις σε συνδυασμό με την εντολή που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών. Θα πρέπει να ακουστούμε πιο πολύ για τα άρθρα τα οποία θα πρέπει να επικυρωθούν. Έχουμε το δικαίωμα της έγκρισης στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά θα πρέπει να συμμετέσχουμε σε πολύ πιο πρώιμο επίπεδο. Κατά δεύτερον, προφανώς θα πρέπει να συζητήσουμε τις συμφωνίες είπα, για τις χώρες ΑΚΕ με πολύ πιο δομημένο τρόπο. Όχι μόνο για τις ίδιες τις συμφωνίες, αλλά και σε συνδυασμό με τις διάφορες διαδικασίες, με τις διάφορες πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα η εργική πολιτική, η εξαγωγή και οι εξαγωγικέ ενισχύσει, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα πακέτο. Και μίλησα με κάποιου ε, πρεσβευτές ε, των χωρών και στην Ρουάντα και θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τρόπου διαπραγματεύσεων. Πώς μιλάμε δηλαδή προς τις χώρες ΑΚΕ, γιατί συχνά έχουν την αίσθηση ότι οι συμφωνίες ΑΚΕ τους επιβάλλονται. Όχι ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια κοινή και αμοιβαία συμφωνία και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Ζαντό. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος ε, Άστον στην προηγούμενη της ε, παρουσία στην Επιτροπή είχε πει σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διτεθειμένη να κάνει πιο ελαστική την εφαρμογή της ρήτρας του πλέον ε, ευνοημένου κράτους για να διευκολύνει κάποιες διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης. Έχει υπάρξει εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Εγώ δεν ήμουν στη Λουάντα, αλλά από ό,τι άκουσα υπήρξε μια έντονη ανησυχία και μια σημαντική δήλωση για την Κοπεχάγη για τη σπουδαιότητα αυτής της διάσκεψης κορυφή, τα προβλήματα της αποψήλωσης, τη ανάγκη υποστήριξη. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη θέληση να συμπεριλάβει και το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές ε, στι Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής σχέση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ε, δασονομικών προϊόντων ή όλα τα εμπορικά στοιχεία που είτε έχουν κάποια επίδραση στην υπερθέρμανση του ε, πλανήτη, είτε το αντίθετο συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υποβάλω και εγώ τις ερωτήσεις μου. Ήσασταν αρκετά ακροθυγείς, αλλά αναφέρατε την συμφωνία με το Καρή Φόρουμ. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τη θέσπιση κάποιων θεσμικών οργάνων με βάση τη Συμφωνία Καριφόρου. Δεν ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις που στείλαμε στη JPA. Μήπως θα μπορούσατε να μας στείλετε το σχετικό κείμενο. Και εις επίρρωση στον νότο όσον είπε ο Ντέιβιτ για την κατάσταση στην Αφρική. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για το κατά πόσο ο Μάιος του 2010 είναι το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση, είναι το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση των βασικών τριών ε, εμπορικών μπλοκ. Πιστεύετε ότι θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα του Μαΐου του 2010. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όσους ε, υπέβαλαν αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Μερικές όμως θα τις αφήσω στον Επίτροπο Ντεχάχτ, γιατί είναι πολιτικής φύσης και καλύτερα να τις ε, συναντήσετε, να τις συζητήσετε με τον αρμόδιο Επίτροπο και όχι με έναν απλό υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο που σας δώσαμε, νομίζω ότι δίνει κάποιες απαντήσεις για κάποιες πληροφορίες που διέρευσαν στον τύπο ότι ε, ήταν τελείως αδρανής η κυρία Άστον και δεν συνέβη τίποτα κατά τη δική της θητεία. Νομίζω ότι το έγγραφο περιλαμβάνει αδιάστατα επιχειρήματα που καταρρύπτουν αυτή τη θέση που εμφανίστηκε σε κάποια άρθρα στον τύπο για την αδράνεια της ε, Επιτρόπου Άστον. Φαντάζομαι είναι μια συζήτηση που θα τη συνεχίσετε είτε με την ίδια την κυρία Άστον είτε με το διάδοχό της. Ο Επίτροπος Δεχάχτ, από ό,τι ξέρω έχει ήδη δώσει κάποιες ενδείξεις για το πώς αντιμετωπίζει τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και θα τις συζητήσετε και στην ακρόασή του. Από ό,τι ξέρω πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρενοχλεί σε καμία περίπτωση τις ε, χώρες ΑΚΕ για τις διαπραγματεύσεις ε, των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης. Θα συνεχιστεί η προσέγγιση της προηγούμενης επιτρόπου στο θέμα αυτό, της κυρίας Άστον. Σε ό,τι φορά τα σχόλια που ανέκυψαν στην μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι οι συμφωνίε οικονομικής εταιρικής σχέσης και η σχετική διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποια θέματα του ανταγωνισμού ή διαφορών ανταγωνιστικότητας. Και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα και μέτρα στήριξης που προσπαθούν να διορθώσουν αυτές τις διαφορές. Επίσης το θέμα των επιδοτούμενων εξαγωγών είναι κάτι πολύ οικείο. Δεν αφορά μόνο τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, γιατί οι χώρε που αναφέρονται δεν εφαρμόζουν ακόμη τέτοιε συμφωνίε τέτοια μέτρα ΕΠΑ. Και σίγουρα οι συμφωνίες και εταιρική σχέσης είναι ένα πλαίσιο για την αναζήτηση μια αμοιβαία εποφελούς ε, λύση, αλλά δεν δημιουργούν τα προβλήματα αυτέ οι συμφωνίε. Σε ό,τι αφορά το θέμα τη ελαστικότητα που εφάρμοσε η επιτροπο Άστον για τη ρήτρα του πλέον ευνο, ευνοημένου κράτους. Η ρήτρα του πλέον ευνοημένου κράτους είναι ρήτρα μη διακριτικής μεταχείρισης. Και τίποτα στη ρήτρα αυτή δεν εμποδίζει ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, ευάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Το αντίθετο. Οι περιοχές με τις οποίες διαπραγματευόμαστε επιφυλάσσονται το δικαίωμα τους ε, να καταλήξουν σε ευνοϊκότερες συμφωνίες ε, μεταξύ τους. Οπότε δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της ρήτας του πλέον ευνοημένου κράτους και της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης παρέχουν και ένα φόρουμ για τη συζήτηση των περιβαλλοντικών μέτρων. Τουλάχιστον αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η διάμεση οικονομική συμφωνία με το Καμερούν επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα δάση και τη δασοκομεία. Ή την μεταχείριση των περιβαλλοντικών αγαθών στα θέματα της απελευθέρωσης. Όλα αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί μόνη της να κινήσει τα πράγματα θέλουμε κάποια προθυμία και βούληση και από τους εταίρους μας για να προχωρήσουμε. Μας ζητήσετε τις ε, πρόσφατες εξελίξεις ότι αφορά την ε, σύστηση θεσμικών οργάνων για το Καριφόρουμ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, εφαρμοστεί τα μέτρα. Θέλουμε σε αρχές του 2010 να πρωτοσυνεδριάσει το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Καραϊβικής, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από την προθυμία των εταίρων μας. Το έγγραφο σε ό,τι αφορά την ε, μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Νομίζω ότι το έγγραφο που σας ε, μοιράσαμε για Τη συνεδρία αυτή είναι πολύ πιο διεξοδικό. Το background paper που σας δώσαμε περιέχει τις τελευταίες εξελίξεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ελάχιστες ήταν ε, μεταγενέστερες εξελίξεις και σας τις επισήμανα. Τέλος, σας χρωστώ και μία απάντηση για το πόσο είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα του Μαΐου του 2010. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ για αυτό το θέμα, δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί πολλές προθεσμίες στο μέλλον αθετήθηκαν. Και για να σας δοθεί μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη θα διαβιβάσω την ερώτηση σε κάποιον πιο αρμόδιο. Όπως είπε και ο Ντέιβιτ, δεν είναι σίγουρο ότι λάβαμε αυτό το background paper που είπατε. Δεν μας το ξαναστένατε καλύτερα, γιατί ίσως χάθηκε κάπου, παράπεσε κάπου και δεν το έχουμε λάβει. Ξαναστείλετε το λοιπόν και εμείς θα φροντίσουμε να το μοιράσουμε στα μέλη της Επιτροπής μας, ο Ντέιβιτ. Καλώς. Να επανέλθω στη ρήτρα του πλέον ευνομένου κράτους. Αυτή δεν ήταν μόνο δήλωση της κυρίας Άστον. Συμφωνήθηκε στην Ολομέλεια ως τμήμα του πακέτου για την αποδοχή της Συμφωνίας Καριφόρουμ. Άλλωστε, δεν είναι θέμα τόσο περιφερειακή ολοκλήρωση. Είναι θέμα ε, οι χώρε του Καριφόρου να μπορούν να συνάπτουν ευνοϊκότερε μεταξύ του συμφωνίε χωρί να, ζητούν τη δική μα ε, σύμφωνη γνώμη. Βέβαια, είπαμε αν το Καριφόρουμ διαπραγματεύεται μια ευνοϊκότερη ρήτρα με τη ΣΥΠΑ, εμεί γιατί να μην αποφεληθούμε. Αλλά αν οι χώρε τη Καραϊβική συνάψουν συμφωνία με τι χώρε τη Αφρικανική Υπήρου θετική για την ανάπτυξη, τότε δεν θα πρέπει αυτόματα να επικαλούμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη ρήτρα του πλέον ευνοημένου κράτους και να διεκδικούμε αντίστοιχη μεταχείριση. Πάντως είναι ακόμη πολύ πρόωρο για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτή η Συμφωνία Καριφόρουμ. Θέλουμε να αρχίσει να λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης για να ενημερωνόμαστε τακτικά για τέτοιου είδους υποθέσεις και να φροντίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, συμφωνεί όχι μόνο αυτή, να εφαρμόζει όχι μόνο αυτή τη συμφωνία, αλλά και οποιασδήποτε άλλες συμφωνίες με το Καριφόρουμ. Όντως, περί αυτού πρόκειται. Δεν θέλουμε να υποστούμε εμείς διακριτική μεταχείριση έναντι των σημαντικότερων μας εμπορικών εταίρων. Πάντω η, χώρα του πλέον, η ρήτρα του πλέον Ευρωπαϊκού κράτου δεν εφαρμόζεται για τι συμφωνίε Καραϊβική Αφρική. Δεν ήταν στόχο τη ρήτρα αυτή να καλύπτει και τέτοιες σχέσει, οπότε ελπίζω να σα καθησυχάζει αυτό. Well, further Αν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι το θέμα αυτό θα συνεχίσει να απασχολεί την Επιτροπή και προφανώς θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε το θέμα αυτό, καθώς και τις δράσεις ε, του καινούργιου επιτρόπου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον Πίτερ Ουάλλας. Πίτερ, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ σήμερα. και που ακούσατε και τα θέματα αυτά σχετικά με τις συμφωνίες είπα, γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσουμε στο σημείο 9 για την 7η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ που έλαβε χώρα στην Γενέβη. Περίπου 300 3.000 ε, ήταν οι αντιπρόσωποι που έλαβαν ε, μέρος και εκπροσωπούσαν 150 χώρες και το ευρύτερο θέμα ήταν φυσικά η τρέχουσα οικονομική κρίση που μαστίζει όλες τις χώρες και οι διαπραγματεύσεις οι Και παράλληλα με την ιδέα των Υπουργών να αναθεωρήσουν το πλαίσιο του ΠΟΗ για να πετύχουμε ένα πολυμερές λειτουργικό εμπορικό σύστημα. Παράλληλα λοιπόν με τις ε, άλλες εκδηλώσεις, τις εργασίες της ΔΟΧΑ και ούτω καθεξής. Πάντα ήταν προσωπική μου άποψη ότι όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική προκειμένου να εξέλθουν των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την οικονομία και το εμπόριο. Πάντα πίστευα στις, ε, στο ελεύθερο, στην ελεύθερη αγορά και θεωρώ ότι το εμπόριο μας ε, δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα τις περιόδους ύφεση. Συμμετείχαμε λοιπόν και εμείς ε, και συναντηθήκαμε με την Πασκαλαμή, την Επιτροπό Άστον, την κυρία Μπέλ, τον ε, Σουηδό Υπουργό Οικονομίας. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής ε, οικονομίας, εκπροσώπους ε, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ε, ευρωπαϊκών συνδικάτων. Και όπως είπα, θεωρώ ότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι πολλές και ότι είναι τεράστιος ο ρόλος τον οποίο θα πρέπει να διαδραματίσει η Επιτροπή μας στο μέλλον. Έχουμε μακρά παράδοση στην Επιτροπή αυτή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές στη Γενέβη. Επτά μέλη του Κοινοβουλίου συμμετείχαν και ξέρω ότι ένας από αυτούς είναι ο Ντάνιελ, ο οποίος και βρίσκεται εδώ, αλλά θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από τον Πίτερ να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Το επόμενο θέμα θα λάβει χώρα και κλεισμένο των θυρών. Πείτε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα ευγενικά σας λόγια. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα και για τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να συναντηθούμε με την Επιτροπή σας και με τους βουλευτές. Και είχα την τιμή να γνωρίσω τους ε, προέδρους, να συναντηθώ με τους προέδρους των Επιτροπών και να κάνουμε καλές συζητήσεις τόπου. Μία ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ήταν καλή η συνάντηση αυτή. Δεν επρόκειτο για μια συνάντηση, όμως την οποία είχαμε οραματιστεί έτσι. Αρχικά θα ήταν πολύ καλύτερο στη σύνοδο αυτή να αποφασιστούν τα πιο σημαντικά στοιχεία για τον γύρο της Δόχας. Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αυτό δεν συνέβη γιατί η τελευταία σοβαρή απόπειρα τον Ιούλιο το 2008 απέτυχε και έτσι ο γύρος της ΔΟΧΑ μάλλον αγκομαχώντας προχωράει παρά με πλήρη ορμή. Υπό τις συνθήκες λοιπόν αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια αξιόπιστη πρόβλεψη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του γύρου της ΔΟΧΑ. Όπως ξέρετε το G20 στο Pittsburgh το επιβεβαίωση των στόχων να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις οι δικές τους μέχρι το 2010 και όλοι το συζήτησαν αυτό, όλοι το έχουν υπόψη τους, αλλά δεν μπόρεσε να ληφθεί σαφής απόφαση. Και άρα το θέμα αυτό δεν ήταν στην επίσημη ημερήσια διάταξη της Συνόδου. Πέραν τούτου, ανέκυψε πολύ συχνά το θέμα αυτό και σε επίπεδο αρχηγών κρατών και είναι σαφές ότι μια συντριπτική πλειοψηφία του ΠΟΕ θέλει να ολοκληρωθούν γρήγορα διαπραγματεύσει βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί ως τώρα για να μην ξαναξεκινήσουν κεφάλαια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι σαφές ότι κάποιοι εμπορικοί εταίροι, κάποιες ε, χώρες δεν είναι έτοιμες να προχωρήσουν, να δώσουν την τελική όθηση, ιδιαίτερα οι ΙΠΑ που θέλουν να γίνουν πιο πολλές συναντήσεις κατηδίαν για να διευκρινιστεί η κατάσταση. Και θα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποια άλλα μέλη του ΠΟΕ, τα οποία και αυτά δεν μπορούσαν να προσυπογράψουν τον Ιούλιο του 2010 το σχετικό πλαίσιο το οποίο είχε κατατεθεί τότε. Συνεχίστηκαν οι εργασίες των εμπρεκνομόνων και πρόσφατα μετά την ανεπίσημη σύνοδο στο Δελχή το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει και διαδικασία διαπραγμάτευση σε υψηλό επίπεδο. Σε δύο εβδομάδε. κατά πάσα πιθανότητα, έχει προγραμματιστεί μάλλον και άλλη συνάντηση και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν και άλλες συναντήσεις και το επόμενο έτος. Όλοι συμφωνούν ότι μέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί τα βασικά πλαίσια μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2010. Γι' αυτό ο Γενικός Διευθυντής Λαμή προβλέπει σοβαρές συναντήσεις μέχρι το Μάρτιο για να αναλύσει το πώς θα έχει εξελιχθεί η κατάσταση ως τότε. Τέλος, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διαδικασία του γύρου της ΔΟΧΑ, Το εμπόριο δεν ήταν αυτό που προκάλεσε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αλλά ενδεχομένως να συμβάλλει τα μάλα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της. Και σε ό,τι αφορά την δημιουργία ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε να υπάρξει πολιτική υποστήριξη και η πολιτική στήριξη αυτή που έχει εκφραστεί πολλές φορές στους τελευταίους μήνες να μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι απόλυτα δεσμευμένη. Η υπουργική διάσκεψη λοιπόν εστιάστηκε σε θέματα τα οποία μπορεί να είναι λιγότερο, αν θέλετε, να τραβούν λιγότερα την προσοχή, αλλά είναι εξίσου σημαντικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΠΟΕ και την αντιμετώπιση των, των τρεχόντων προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά την Ντόχα υπάρχει μια σημαντική ανησυχία, το να συμβεί δηλαδή μια επαναχώρηση ό,τι αφορά την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών. Ήδη δυσχερής οικονομική κατάσταση έχει ήδη, για παράδειγμα, ε, χειροτρέψει την κατάσταση σε αρκετές χώρες. Κάποιες χώρες όπως η Ρωσία, και οι Αργεντινοί αποτελούν την εξαίρεση, γιατί οι πιο πολλές άλλες χώρες δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ε, αναστροφής της απελευθέρωσης της αγοράς. Ελπίζουμε αυτό να παραμείνει έτσι. Ο ΠΟΕ έχει συστήσει ένα σχετικό μηχανισμό εποπτείας για να υπάρξει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά και που αποτελεί μια ευκαιρία για να συζητούνται τέτοια θέματα. Και τέλος, η εποπτική αυτή δραστηριότητα αποτελεί και ένα είδος, αν θέλετε, ε, πηγής πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις στα διεθνή φόρα. Και σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια του G20. Άρα, από αυτή την άποψη ήταν σημαντική η σύμβολη της υπουργικής διάσκεψης σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του εποπτικού μηχανισμού, τονίζοντας ε, την ανάγκη να δίνονται από τα μέλη του ΠΟΕ πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται. Επίσης υπήρχαν και κάποιοι άλλοι τομείς που συζητήθηκαν, όπου έχει σημειωθεί και έχει προταθεί μάλλον πρόεδρος. Καταρχάς για την ενίσχυση των μηχανισμών αναθεώρησης της εμπορικής λειτουργίας. Πρόκειται για ένα φόρουμ μεταξύ ομοτήμων, όπου οι χώρες ΠΟΕ μπορούν να εξετάζουν η μία τα μέτρα που έχει επιβάλει άλλα και να συζητούν τα μέτρα αυτά. Στα πλαίσια του εμπορικού των εμπορικών πολιτικών. Επίσης έγιναν συζητήσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και πάλι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πολύ ένθερμα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την κατάρτιση των νόμων είναι πολύ διαφανές. Έγινε επίσης μια συζήτηση για τον ρόλο των περιφερειακών ε, εμπορικών συμφωνιών, των ε, προνομιακών συμφωνιών και το πώς θα μπορούν να, να διαμορφώνονται προκειμένου να μην υπονομεύουν αλλά να ενισχύουν την απελευθέρωση της αγοράς. Συνολικά λοιπόν ήταν πολύ εποφελής στη συνάντηση αυτή, όχι επειδή συμπεριλήφθηκαν τα απαστράπτοντα αν θέλετε θέματα τα οποία ελπίζαμε να συμπεριληφθούν, αλλά διαπιστώσαμε ότι τελικά αυτό ήταν το καλύτερο περιεχόμενο σε ό,τι αφορά την υπουργική διάσκεψη. Ευχαριστώ, Πίτερ, λέει ο Πρόεδρο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που παραβρέθηκε εδώ σήμερα. Είσαι από τα πολύ συνεπή μέλη εδώ στην Επιτροπή μας και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής. Ξέρω ότι και ο Ντάνιελ ήταν παρόν, αλλά να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ. Εγώ δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στην Υπουργική Διάσκεψη, γιατί η αντιπροσωπεία ήταν μόνο επταμελής και δεν χωρούσε και εκπρόσωπος της δικής μου ομάδας. Εντάξει, δεν τα έβαψα και μαύρα, ειδικά μετά από αυτά που μας εξηγήσατε για την ε, διάσκεψη αυτή. Και μάλιστα διαβάζοντας ε, τη σύνοψη του Προέδρου που μας μοιράσατε, δεν έχω την αίσθηση ότι ε, ήταν πολύ καρποφόρα συνεδρίαση. Έγινε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, αλλά καμία σχεδόν συμφωνία. Ήταν πραγματικά πολύ αφηρημένη η συζήτηση και τελείως διασπασμένη. Στη σύνοψη του Πρόεδρου υπάρχει αυτή η ιδέα ότι συμφωνούμε να μην ξανανοίξει συζήτηση για συμπεφωνηθέντα ζητήματα. Κάτι που δεν φαίνεται να εστερνίζεται ο Αμερικανός συνομιλητής, ο κύριος Κέρκ. Εσείς με ιδιαίτερο ενθουσιασμό μας δώσετε ραντεβού στην επόμενη υπουργική διάσκεψη ε, για να υλοποιηθεί, για να ολοκληρωθεί ο γύρος της ε, Ντόχα. Εγώ έχω απελπιστεί ότι δεν πρόκειται να ε, κερδίσει η ομάδα η Εθνική Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εσείς τι, πού στηρίζετε τις ελπίδες σας ότι θα ολοκληρωθεί επιτέλους την επόμενη φορά ο γύρος της Ντόχα. Γιατί έχουμε πολλές νέες εμπορικές προκλήσεις. Χρηματοπιστωτική κρίση, οικονομική κρίση, νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις, νέες κοινωνικές προκλήσεις. Και κάποιες προκλήσεις που σχετίζονται με τη σύναψη άλλων διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Παρ' όλα αυτά πιστεύετε ότι θα διεκπαιρεωθεί κάποια στιγμή ο γύρος της Ντόχα ή μήπω είναι η ώρα επιτέλους η Ευρώπη να σκεφτεί είτε να προτείνει μια αναθεώρηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου ή τουλάχιστον να αλλάξει το πρόγραμμα των διαπραγματεύσεών της στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ώστε να επανέλθει η πολυμερής εμπορική διαπραγμάτευση στη σύγχρονη εποχή και να εγκληματιστεί με τις νέες εξέλιξεις ο κύριος Τούρακ. Ευχαριστώ συνάδελφε πρόεδρε. Ως ε, πρώην μέλος συμμετείχα στην αντιπροσωπεία και θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ημέρα της Λισαβόνας, την πρώτη μέρα δηλαδή που τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Και μου δόθηκε η εντύπωση ότι στον ΠΟΕ παρακολουθείται με ακρίβεια το γεγονός ότι πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά. Αλλά το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο βρισκόμαστε σε ίδιο επίπεδο όντω με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή μας στο Συμβούλιο. γιατί υπάρχει κάποια, α, κάποιο προβάδισμα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που έχει το Συμβούλιο. Εμείς εξαρτώμαστε από την Επιτροπή. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Θα πρέπει αυτό να το συζητήσουμε πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά δεύτερον, η εντύπωση που δόθηκε σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της Επιτρόπου Μαριάν Φίσερ η οποία και πάλι δήλωσε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα. Και ότι υπάρχει πάντα το ερώτημα του κατά πόσο υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση. Τέθηκαν λοιπόν τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος μας είπε ότι συχνά ακούγονται και επικρίσεις στα πλαίσια της ε, Συνόδου, κυρίως από την Αμερική αλλά και από άλλους. Και ο εκπρόσωπος τον ΗΠΑ είπε ότι θα έπρεπε να κάνουν και μεγαλύτερες προσφορές και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα θα καταφέρουμε όντω τους επομενους τρεις τρεις-τέσσερις μήνες να δώσουμε μια τέτοια όθηση στον κύριο της Δόχα ή θα πούμε ότι παρατούμαστε γιατί δεν μπορούμε φυσικά να παρατηθούμε από τώρα. Θα ήταν λάθο αυτό. Θεωρώ ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλουμε προκειμένου ο γύρος της Ντόχα να λάβει καινούρια όθηση, να υπάρχει πολιτική θέληση. Θα πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό, θα πρέπει να το αποπειραθούμε. Γιατί πάντα είναι καλύτερε οι πολυμερεί από τις διμερείς συμφωνίες. Ρωτώ λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει, αν θέλετε, το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις τρέχουσες προτάσεις ή και υπερβαίνοντας τις τρέχουσες προτάσεις θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά τις είπαμε τους άλλους εταίρους προκειμένου να πετύχουμε συμφωνία το 2010. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Όχι να πούμε, όπως είπε ο συνάδελφος Ζαντό, ότι... Να πούμε, όπως είπε ο συνάδελφος Ζαντό, ότι είναι ούτως ή άλλως καταδικασμένος ο γύρος της Δόχα. Ευχαριστώ. Δεν, ξέρω αν είναι εύκολο αυτό το να παίξουμε το διαμεσοβουλευτικό ρόλο με τη ΣΥΠΑ. Ο Ντάνιελ συνάδελφοι. Και εγώ είχα την τιμή να συμμετάσχω στη Γενέβη και μου φαίνεται ότι στα πλαίσια της Δόχα δεν προχώρησε τίποτα, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο και να εξαγάγω το εξής συμπέρασμα. Θυμάμαι πολύ καλά το πρώτο μου ταξίδι στα πλαίσια συνάντησης του ΠΟΕ στο Χονγκ Βρεθήκαμε λοιπόν στο Χονγκ Κόνγκ μία εβδομάδα και θυμάμαι ότι καθημερινά υπήρξε ενημέρωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς είχαν οι εξελίξεις οι διαπραγματευτικές. Και ξέρω ότι ήταν πολύ δημοφιλής ε, η ενημέρωση αυτή και μας ζητούσαν να συμμετάσχουμε κι εμείς για να ενημερώνονται όλοι από πρώτο χέρι. Αυτό λοιπόν το 2005. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πάρουμε ως υπόδειγμα. Όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά για να ακολουθούμε από κοινού κοινέ στρατηγικές. Να υπενθυμίσω ότι έγιναν συζητήσεις με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις, το οποίο είναι και θετικό, αλλά τελικά ήταν κοινοί οι στόχοι, κοινέ οι στρατηγικές και έτσι είχαμε τη δυνατότητα στις συζητήσεις με βουλευτές και από άλλες χώρες με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, με εκπροσώπους ενώσεων και επαγγελματικών συνδικάτων, να παρουσιάσουμε μια ενιαία στάση και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πόσο μάλλον τώρα που έχει τεθεί και σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Να είναι κοινέ δηλαδή η κοινή στάση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε μέχρι την επόμενη συνάντηση στα πλαίσια του ΠΟΕ. Προκειμένου να διατυπώνουμε δηλαδή τις ίδιες απόψε απόψεις. Αυτό θα πρέπει να είναι το δίδαγμα της Γενέβης. Γιατί τα πράγματα από αυτή την άποψη δεν πήγαν και πολύ καλά στη Γενέβη. Και από πλευρά Κοινοβουλίου και από πλευρά Επιτροπή. Εάν δεν υπάρχουν ε, σημεία, θα ήθελα να πω αυτά που είπε και ο Ντάνιελ. Μετά από την επίσκεψη στο Χονγκ Κόνγκ είχαμε μια πολύ καλή ενημέρωση, όχι από την ε, Γενική Διεύθυνση μόνο εμπορίου αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας που είχε πάει στη συνάντηση αυτή. Το θέμα των σχέσεων τώρα με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πριν λίγο καιρό συζητήσαμε ποια είναι τα προβλήματα με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είχα και εγώ μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη και άλλους εκπροσώπους και υπάρχει η αίσθηση και είναι σαφής η αίσθηση αυτή ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή τη φάση έχουν τόσα εσωτερικά προβλήματα, ε, γίνεται πιο σημαντικό το γεωργικό λόμπι. Ο Πέτερ Μάντελσον προσπάθησε να σπάσει το αδιέξοδο στα πλαίσια της συζήτηση για τη γεωργία. Διαρωτώ με αν αυτό τώρα έχει ξαναοδηγηθεί στο προηγούμενο επίπεδο και αν οι Αμερικανοί έχουν ξαναγίνει πιο κλειστοί και πιο προστατευτικοί Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. που δείχνουν και τη σωστή συνεργασία του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη στενή συνεργασία και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα περισσότερα από τα σχόλια έχουν ένα κοινό θέμα θα έλεγα Καταρχάς πρέπει να πιστεύουμε πάντα στην Τόχα και αν ναι, τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε με την Τόχα. Μετά από τόσες περιτές, περιτούς συναγερμούς θα έλεγα, ίσως να έχουμε χάσει στη διαδικασία ενώ κάποια από την αξιοπιστία της και να μπορέσουμε να τερματίσουμε τη διαδικασία αυτή όπως αποτύχαμε και τον προηγούμενο Ιούλιο. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα ιστορικό προηγούμενο παρηγορητικό. Στα πλαίσια της ιστορίας του Γκάτ, κανένας γύρος δεν έκλεισε εγκαίρος. Μέχρι τώρα κανένας δεν είχε αποτύχει επίσης. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και η Ντόχα δεν θα είναι η εξαίρεση. Ένα άλλο ιστορικό παράλληλο στοιχείο είναι ο γύρος της Ουρουάης. Κράτησε 8 χρόνια. Και το γάτε εκείνη την εποχή είχε 120 μέλη. Τώρα έχουμε 153 μέλη στα πλαίσια του ΠΟΕ. Εκπροσωπούνται πολύ περισσότερες κατηγορίες χωρών και συμφερόντων και είναι μια οργάνωση ο ΠΟΕ που δουλεύει στη βάση της συνένεσης και έτσι το μικρότερο μέλος του ΠΟΕ έχει ουσιαστικά ένα de facto δικαίωμα βέτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να καταλήξει κανείς σε συμβιβασμούς ανάμεσα στις χώρες αυτές. από τις λιγότερο αναπτυγμένες μέχρι τις πιο πλούσιες. Και αυτό εξηγεί θα έλεγα τις καθυστερήσεις που έχουν προκληθεί. Παραμένουμε αισιόδοξοι όμως, είναι εφικτή η επιτυχία και ελπίζω να την πετύχουμε στο μέλλον. Αναφερθήκατε όλοι στον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το 2008, όταν πράγματι είχε φανεί ότι τερματίζαμε τη διαδικασία, και η ΙΠΑ από τη μία και η Ινδία και άλλες χώρες από την άλλη ήταν η αιτία που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις. Η νέα κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πράγματα στη ΣΥΠΑ είναι πραγματικά ενδιαφερόμενη για να προχωρήσει στην εμβάθυνση των σχέσεων με άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας θα φανεί και στα πλαίσια του ΠΟΕ. Είναι βέβαια σαφές ότι τον πρώτο χρόνο του ο πρόεδρος Ομπάμα είχε άλλες κατεπίγουσες θα έλεγα προτεραιότητες το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών, την Κοπενχάγη και μέχρι τώρα δεν στάθηκε ικανός να συγκεντρώσει την προσοχή του και να αναλάβει τις προσπάθειες που απαιτούνται στις διαπραγματεύσεις για την Τόχα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει ένας έντονος σκεπτικισμός για το γύρο της Ντόχα και για τα αποτελέσματα στα οποία έχουμε μέχρι τώρα καταλήξει. Ο επιχειρηματικός κόσμος και όχι μόνο η γεωργία, αλλά και ο βιομηχανικός γενικά τομέας και λιγότερο οι υπηρεσίες, αλλά τα δύο αγαθά, γεωργία και βιομηχανία δηλαδή, προϊόντα, θεωρούν ότι έχουν ε, υποχωρήσει σε πολλά και έχουν κερδίσει λίγα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε αναζητούν τρόπους να δούνε ακριβώς ότι περαιτέρω προσβάσει σε αγορές μπορεί να πετύχουν από τις τρεις χώρες στόχου Βραζιλία, Ινδία και Κίνα. Αυτό τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα για τα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και για τα γεωργικά. Συνεχίζουν διμερείς διαπραγματεύσεις με αυτές τις τρεις χώρες. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, αν και όχι συνολική. Τώρα θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο γεφυροποιού. Προσπαθούμε. Το πετύχαμε μέχρι τον Ιούλιο, ιδιαίτερα στη Γεωργία, βοηθήσαμε να υπάρξει μια συνένεση στο πιο προβληματικό τομέα, τις ειδικέ ρήτρες προστασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά σε αυτή τη φάση υπάρχουν ε, γενικά σοβαρές διαφορές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές τους και δεν θα πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να πληρώνουν γι' αυτό και για χώρες όπως η Αργεντινή και η Νότιος Αφρική έχουν, ε, θεωρούν οι ΙΠΑ ότι έχουν ε, δώσει πάρα πολλά προς τις χώρες αυτές και ε, θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει και υπέρ των ΙΠΑ η σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ρόλος μας συστηματικά το να αναζητούμε να παίξουμε το ρόλο του γεφυροποιού, αλλά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ήμασταν κινητήρια δύναμη αυτής της διαδικασίας εδώ και χρόνια. Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία συνάντηση. Και πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση όταν η κυβέρνηση τον είπα και ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να ρίξει το βάρος του στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης και αυτό θα πιέσει και τις υπόλοιπες χώρες του ΠΟΕ. Δεν θα καθυστερήσει νομίζουμε πολύ η στιγμή αυτή. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τα προσυζήτηση θέματα προς τον ΠΟΕ για να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση ή διαπραγματεύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό τώρα και για λόγους ουσίας και για λόγους πολιτικούς. Καταρχάς κανείς δεν είναι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος να εγκαταλείψει την Τόχα παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν. Καμία χώρα από τους ομιλητές στην Υπουργική Συνάντηση ή σε άλλα επίπεδα δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει την Τόχα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήθελε κανείς να πάρει ένα τόσο αντιλαϊκό μέτρο. Και σε επίπεδο ουσίας η φιλελευθερωποίηση του εμπορίου, των αγαθών και των υπηρεσιών στην ουσία προετοιμάζει θα έλεγα το έδαφος για άλλες συμφωνίες σε άλλες δραστηριότητες και τομείς του ΠΟΕ αν δεν ε, πετύχουμε σημαντικά βήματα προόδου στα συγκεκριμένους τομείς, τι θα μπορούσε να ελπίζει κανείς ότι θα πετύχει ε, στα υπόλοιπα πλαίσια του ΠΟΕ, που δεν έχουν καν τεθεί σε συζήτηση αυτή τη στιγμή, όπως οι επενδύσεις, οι δημόσιες προμήθειες, τα θέματα του περιβάλλοντος ή τα θέματα της εργασίας Αυτά τα θέματα είναι βέβαια θέματα που αποκλείουν οι περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο βασικό ρόλο του ΠΟΕ, την απελευθέρωση δηλαδή των υπηρεσιών και των αγαθών και να βοηθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή των διεθνών συμφωνημένων κανόνων και δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική δυνατότητα στο να αποστρέψουμε την προσοχή μας από και εμείς και οι αναπτυσσόμενες χώρες προς άλλες κατευθύνσεις από την Τόχα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, θα εμείνουμε στα πλαίσια της Ντόχα και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες παράλληλα Υπάρχει το θέμα των προτιμησιακών συμφωνιών της Ένωσης με άλλες συμφωνίες, με άλλες ομάδες μάλλον και χώρες του ΠΟΕ. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα μπορεί να προχωρήσει, αλλά υπόκειται και στην πρόοδο των πολυμερών απελευθερώσεων τομέων. Για την καλή συνεργασία τώρα ανάμεσά μας και, και στο Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, Έχουμε τώρα έναν προσωρινό επίτροπο για μία περίεδο προσωρινή, την κυρία Μπενίτα Φερέρο Βάλνερ, η οποία παραμένει επίτροπος μέχρι το τέλος ισχύω αυτής της επιτροπής. Συνεργαζόμαστε με τη Φερέρο Βάλνα, συνεργαζόμαστε και με τον Κάρελ Ντεχούχτ, και όπως και με τους προκατόχους τους θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε περαιτέρω την καλή αυτή σχέση τη διοργανική. Όπως το προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τομείς συνεργασίας σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, Σαν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε να συνεργαζόμαστε και να σας δίνουμε ό,τι στοιχεία απαιτείτε. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο γύρω από αυτά που είπατε για τη ΣΥΠΑ. Πρώτον, αναφερθήκατε στις διαπραγματεύσεις ότι παραχωρούν πολλά. Πάντα το λέει αυτό ένας καλός διαπραγματευτής για να κατηγορήσει το διαπραγματευτή του. Όταν παλαιότερα είχα εμπλακεί με την ένωσή μου ε, σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, θυμάμαι στα πλαίσια του γύρου της Ουρουάης ότι είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ, είπα. Και είχαμε χαρεί πολύ ότι τους ε, είδαμε γύρω από την τράπεζα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει στη συμφωνία του Blair House, άσχετη βέβαια με τον Τόνι Μπλερ. Λοιπόν, η επόμενη συνάντηση, το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ τα μέλη να παραμείνουν. Συντονιστές, βουλευτές, γραμματεία των, της Επιτροπής Επίσημη των Πολιτικών Ομάδων, νομική υπηρεσία. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Να πω επίσης ότι ο Αμερικανός πρέσβης πήρε τα διαπιστευτήριά του και καλό θα είναι η γραμματεία μας να τον προσκαλέσει σε μια συνάντησή μας. Στις αρχές του 10 θα υπάρξει και μία επίσκεψη στη Βραζιλία και γι' αυτό θα πρέπει να προσκαλέσουμε και τον πρέσβη της Βραζιλίας σε μια από τις συναντήσεις μας.